Se Ησυχία σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Σήμερα ξεκινάμε ένα κονκλάβιο που αρχίζει σήμερα και θα τελειώσει όταν θα έχουμε ολοκληρώσει την ψηφοφορία σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, αύριο το βράδυ, μεθαύριο το πρωί, μεθαύριο το βράδυ, τέλος πάντων πριν τις 31 Δεκεμβρίου. Είδατε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής μας, η οποία είναι αφιερωμένη ουσιαστικά στην ψηφοφορία του προϋπολογισμού, στο σχέδιο προϋπολογισμού 2013. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Έχουμε όλες τις γλώσσες παρούσες, αυτά είναι οι ανακοινώσεις του Προέδρου. Εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 6ης Ενάτου. Άμα δεν έχετε παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται οριστικά. Και πάμε στην ψηφοφορία των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού 2013. Σας το λέω ήδη από τώρα. Ο καθένας έχει την, έχετε όλοι δηλαδή την κάρτα ψήφου. Θα έχουμε από ό,τι φαίνεται πολλές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Επίσης, ο κάθε συντονιστής <coughs> να σιγουρευτεί ότι όλα τα μέλη του και αναπληρωματικοί είναι εδώ. Να βλέπω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει την κάρτα ψήφου. Θα λυθεί όμως το πρόβλημα. Αν ο ίδιος συντονιστής ε, μου πει ότι έχω δικαίωμα ψήφου, τότε και εγώ θα το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, τα βασικά μας έγγραφα. Που είναι το κείμενο που έχει και νομική βάση είναι αυτό, αυτή, αυτή η μπροσούρα το έγγραφο αριθμός 4. Θα ήταν πιο απλό να το είχαμε ονομάσει 1, αλλά το ονομάσαμε 4. Θα μου πείτε γιατί θα ήταν πιο απλό. Επίσης, έχετε σε στην την προσούρα αριθμός 4 μόνο νούμερα. Έχετε άλλα 4 τετράδια με τα σχόλια. Θα ψηφίσουμε εμείς ορισμένα από αυτά, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία ευθύς εξ αρχής, αλλά να ξέρετε ότι αυτά αποτελούν τη βάση. Μετά, έχουμε μερικά φέιβολον τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την ψηφοφορία. Ψηφοφορία unblock. Ξέρετε ότι ψηφίζουμε unblock σε πολλές εκθέσεις και φυσικά και για τον προϋπολογισμό. Όταν έχουμε τη συμφωνία των συντονιστών για να ψηφίσουμε unblock, τότε θα ψηφίσουμε unblock. Στα έγγραφα που σας μοιράστηκαν, λείπει ο πίνακας για τα σχέδια πιλότο και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Η γραμματεία. Γράφει αυτή τη στιγμή, συγγράφει μάλλον αυτή τη στιγμή, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν ο εισηγητής με τους συντονιστές. Προτείνω να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν, στο Γενικό Διευθυντή που είναι παρόν. Η Κομισιόν, σύμφωνα με την παράδοση, θα μας θυμίσει τους στόχους και τις γενικές γραμμές του προϋπολογισμού θα μας πει τη γνώμη της για την ψηφοφορία που μεσολάβησε φέτος το καλοκαίρι στο Συμβούλιο Υπουργών, ο εισηγητής θα μας πει πώς προετοίμασε την ψηφοφορία μαζί με τους συντονιστές και μετά θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω τη γνώμη της Κομισιόν μετά από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο και πριν από την ψηφοφορία των τροπολογιών που κατετέθηκαν. Το πρώτο σημείο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι πολλές, με ικανοποίηση πολλές από τις τροπολογίες που κατέθεσε το Κοινοβούλιο αποκαθιστά τις πιστώσεις πληρωμών και υποχρεώσεων που είχε περικόψει το Συμβούλιο κατά την ανάγνωσή του. Οι τροπολογίες αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα κοινό όραμα μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου για το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από παλαιότερες δημοσιονομικές αποφάσεις. Το μέγεθος των περικοπών του Συμβουλίου 5,3 δις ευρώ είναι αβάσταχτο, διότι έκοψε υπερβολικά και για τρίτη συνεχή χρονιά πολιτικές οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο της στρατηγικής 2020 για τις επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Πρόκειται για προγράμματα υπό τον τίτλο 1 ή για την πολιτική συνοχή 1β. Αυτές οι δαπάνες είναι πιο χρήσιμες από ποτέ σε αυτή την περίοδο κρίσης. Και είναι ακατανόητη και η περικοπή του τίτλου, στον τίτλο 4, όπου προτείνει έναν προϋπολογισμό για το 2013, έναν προϋπολογισμό μικρότερο κατά 600 εκατομμύρια ευρώ από την εκτέλεση του 2011. Για τις πιστώσεις πληρωμών είχαμε μία τρίμερη στις 26 Σεπτεμβρίου, πολύ χρήσιμη. Και αυτή η συνεδρίαση τόνισε ότι η Κομισιόν, απέδειξε μάλλον ότι η Κομισιόν με λογική και συγκράτηση αντιμετώπιζε τις δαπάνες. Και Ο προπολογισμό 2013 συντάχθηκε με την εντύπωση ότι εκείνος του 2012 θα <coughs> είχε καλύψει εκείνον του 2012 για τις τροπολογίες που τονίζουν τη θέση του Κοινοβουλίου για τις πιστώσεις πληρωμών, εγώ θα αναφέρω τους ειδικού προσανατολισμούς για τα προγράμματα και δράσεις υπέρ της ανάπτυξης στα πλαίσια του U20 για το e-learning, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Λαβία και τις ειδικέ επιτροπές που έθεσαν και τις γραμμές εκείνες ε, για τη διοικητική υποστήριξη του κάθε προγράμματος που είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία τους. Για μια ακόμη φορά η Κομισιόν απέδειξε ιδιαίτερη συγκράτηση στο σχέδιο προϋπολογισμού και οι περικοπές του Συμβουλίου διακυβεύουν τις δυνατότητες δράσης του θεσμικού οργάνου και της εφαρμογή των προγραμμάτων. Για για τα αποθεματικά σχετικά με τα προγράμματα του τίτλου 1β και του τίτλου 2. Εμείς καταλαβαίνουμε την πολιτική εμβέλεια ορισμένων τροπολογιών, αλλά είναι ουσιαστικό να μην προσθέσουμε ένα στοιχείο δυσδιαχειρισιμότητας σε ορισμένες γραμμές. Εκφράζω επιφυλάξεις για ορισμένα ειδικά ντοσιέ και τη συνεχή πληροφόρηση που πρέπει να δίνει η Κομισιόν για αυτά. Σύστημα ICS2. Αναγνωρίζοντας πλήρως την νομιμότητα και την αναγκαιότητα μιας τακτικής και ακριβούς ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για, την, για το πώς προχωράει αυτό το σύστημα. Εμείς θεωρούμε ότι το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα για το SAS2 είναι ήδη πολύ καλά αποφασισμένα και η Κομισιόν θα συνεχίσει να στέλνει με διαφάνεια και ακρίβεια όλες τις πληροφορίες στο Κοινοβούλιο. Αναρωτιέμαι όμως αν αυτού του είδους μία ε, θέση αποθεματικό έχει, έχει σήμερα νόημα η Κομισιόν σας έχει στείλει μία προσωρινή λίστα από το φθινόπωρο για τα πιλωτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που ελπίζουμε να σας βοηθήσουν. Για να ολοκληρώνω, Πρόεδρε, θέλω να αναφέρω ότι όπως κάθε χρόνο η Κομισιόν προετοιμάζει την επιστολή εξ, εκτελεσιμότητας και θα συνεισφέρει στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής με τις απαραίτητες πληροφορίες. και αναφέρονται εκεί και οι δυσκολίες εκτέλεσης ορισμένων τροπολογιών. Λοιπόν, περιμένω τη συνέχεια των εργασιών. Ε, Ευχαριστώ. Ο εισηγητής τώρα. Να μας εξηγήσει οι συγκητές μάλλον σε τι κλίμα μέσα ετοίμασαν με τους συντονιστές την ψηφοφορία αυτή. Δεν μιλάμε πια για την ουσία, διότι για την ουσία έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Περνάμε στην ε, ψηφοφορία. Αλλά επειδή έτσι κι πρόκειται για την εξέταση 1500 τροπολογιών, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να οργανώσουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, Τζοβάνι, μπορείς να μας πεις λίγο πώς προτείνεις να δουλέψουμε σήμερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ψηφοφορία του, του προπολογισμού είναι πάντοτε ιδιαίτερα πολύπλοκη. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πόσο πολύπλοκη είναι η ψηφοφορία για να έχουμε στο τέλος ένα αποδεκτό αποτέλεσμα. Και το πώς φυσικά αυτό είναι συμβατό με τις στρατηγικές του Κοινοβουλίου. Εμείς ως Κοινοβούλιο θελήσαμε να υπογραμμίσουμε τι σημασία που οι πιστώσεις πληρωμών θα έχουν για το 2013 και αυτό εν ώψη των δημοσιονομικών προοπτικών. Εμείς ε, σε αυτή την Επιτροπή καταφέραμε να πετύχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία που θα μπορέσει να υποστηρίξει τη στρατηγική του εισηγητή. Έχουμε μερικές ε, διστάμενες απόψεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων σχετικά με ορισμένους τομείς και όχι τίτλους, αλλά ελπίζω ότι θα τις ξεπεράσουμε. Προτείνω λοιπόν, Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία από το τέλος. Δηλαδή, να ψηφίσουμε πρώτα τις διοικητικές γραμμές Ξεκινώντας δηλαδή, έχετε τις λίστες ψηφοφορίες. Να ξεκινήσουμε από τις ε, διοικητικές, ε, από τους διοικητικούς καταλόγους ψηφοφορίες, μετά πάμε στις αποκεντρωμένα όργανα και μετά πάμε στο leading 5, leading 3 και 2. Και μετά θα δούμε πού είμαστε, πώς έχουμε προχωρήσει και θα δούμε αν θα συνεχίσουμε σήμερα ή να ψηφίσουμε και θα συνεχίσουμε από το πρωί. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ντέρεκ, έχετε κάτι να προσθέσετε. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ναι. Όπως είπε και ο κύριος εισηγητής, θα δούμε σήμερα τις διοικητικές γραμμές και αύριο προτείνουμε να ψηφίσουμε το Κοινοβούλιο και τα άλλα τμήματα. Οι συνάδελφοι ξέρουν τι συμφωνία έχουμε πετύχει με τις τροπολογίες. Αύριο θα σας προτείνουμε κάποιες προφορίες να γίνουν on block. Θα ψηφίσουμε αύριο και τους προπολογισμούς των άλλων θεσμικών οργάνων, ελπίζω επίσης on block, όλα μαζί δηλαδή. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε. Συνεπώς, καταλάβατε όλοι με ποια σειρά θα ψηφίσουμε τις διάφορες κατηγορίες, έτσι. Θα αρχίσουμε με τις προφορίες οριζόντιου χαρακτήρα για τις διοικητικές γραμμές και τους οργανισμούς και μετά θα πάρουμε την κατηγορία 5 που είναι οι διοικητικές δαπάνες αλλά μόνο τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την κατηγορία 3 α και 3β και την 2, Γεωργία. Και στη συνέχεια θα δούμε που θα έχουμε φτάσει και θα πούμε τι θα κάνουμε μετά. Αύριο το πρωί θα δούμε τους προπολογισμούς των άλλων θεσμικών οργάνων και τις άλλες κατηγορίες, ιδιαίτερα την 1α και την 4, που είναι οι κατηγορίες για τις οποίες έχουμε και τις ε, μεγαλύτερες αποκλίσεις. Οπότε η ψηφοφορία μπορεί να καταλήξει αλλιώς. Σύμφωνοι. Καλώς. Ωραία. Για τις διοικητικές γραμμές πρώτα. Έχουμε τον ε, πίνακα αυτόν. Ο πίνακας αυτός λέει Rapporteur Strategy Administrative Lines 0104 και 0105. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε αμπλόκ, τον πίνακα αυτόν. Όλο τον πίνακα. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Τρεις κατά. Αποχές. Καμία. Εγκρίνεται. Συνεπώς, όλες οι τροπολογίες που έχουν να κάνουν με αυτές τις γραμμές καταπίπτουν, έτσι, γι' αυτό και ψηφίσαμε on block. Έρχομαι τώρα στους οργανισμούς, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Μπορούμε και εδώ να ψηφίσουμε on block. Μαζί δηλαδή όλα. Παρακαλώ κύριε Σιγητά. Μπορούμε να ψηφίσουμε μπλοκ τα νούμερα και μετά έχουμε άλλες μεμονωμένες ψηφοφορίες που πρέπει να γίνουν. Αποκλείονται οι οργανισμοί εποπτείας, δημοσιονομικής υποπτείας. Θα τους δούμε μετά. Καλώς. Ωραία. Ψηφίζουμε όλα μαζί, χωρίς όμως να συμπεριλάβουμε τους τρεις οργανισμούς δημοσιονομικής εποπτείας που θα εξετάσουμε με την γραμμή 1α. Την κατηγορία, διορθώνει ο Πρόεδρος, 1α και κάποια σχόλια τα οποία ίσως ψηφίσουμε χωριστά. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Τέσσερι. Αποχέ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Για τους οργανισμούς λοιπόν έχουμε κάποιες παρατηρήσεις έτσι, και κάποιες επιφυλάξεις. Είναι στο τέλος του ίδιου αυτού πίνακα. Η πρώτη γραμμή είναι μια τροπολογία που έχει αποσυρθεί. Η δεύτερη είναι μια τεχνική τροπολογία που δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Η τρίτη στην κατηγορία 2 επιφύλαξη για αποθεματικό 10% εξαιτία θεμάτων απαλλαγή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ωραία, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Μου λένε όμως ότι εγώ δεν δικαιούμαι να ψηφίσω. Ψηφίστε παρακαλώ. Να επαληθεύσουμε κιόλα αν είναι σωστές οι ψήφοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Στη συνέχεια, περνάμε στο 3α, Frontex. Για την Εροσούρ. Φυσικτή είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια πάτε για τη Frontex έχουμε 75% στο Σέγγεν. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το αποθεματικό μπορούμε να ψηφίσουμε επί της αρχής για τα υπόλοιπα ε, που έχουν να κάνουν με το Σέγγεν και που ανταποκρίνονται στην ίδια φιλοσοφία, τα άλλα 75%. Ποιοι είναι υπέρ. Πάντα για τους οργανισμούς μιλάμε, έτσι, ναι. Και φιλελεύθεροι, ρωτά ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Οι μεγάλες ομάδες, οι πράσινοι και δεύτεροι. Αποχές Ωραία, συνεπώς συστηματικά απορρίπτονται τα αποθεματικά αυτά. Για τη Frontex όμως έχουμε ένα σχόλιο για την Eurosur. Υπέρ, εισηγήτης υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε μας μένει μόνο. Παρακαλώ κύριε Σίγδα. Πρόεδρε, εδώ ξεχάσαμε να ψηφίσουμε κάτι. Ψηφίσουμε για το προηγούμενο αποθεματικό της ΛΥΜΠΕ. 5-6-2-0. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Πρόκειται για τη διάσωση στη θάλασσα. Είναι κατά ο εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται λοιπόν αυτό το σχόλιο. Μας μένει στη σελίδα αυτή τι ακόμα. η τροπολογία της Επιτροπής ΕΝΒΗ με χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα να επανέλθει το σχέδιο προπολογισμού. Αυτό προτείνει ο συγκητής. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ο συγκητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ, κύριε Σιγητά, είναι σε μειοψηφία οι σοσιαλιστές. Άλλη μια ψηφοφορία ξεχάσαμε. Την πρώτη του τίτλου του 5, του τομέα 5, 3551. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν ε, έχω πάρει ακόμα το ρυθμό μου, αυτό φταίει. Λοιπόν, υπάρχει τροπολογία της Utah Hawk που, κακός, ξέχασα. Κατά ο εισηγητής. Ποιο είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή η τροπολογία. Ωραία, τώρα τελειώσαμε με στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Περνάμε συνεπώς στην κατηγορία 5. Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε πρέπει να πάρετε στα χέρια σας ένα φύλλο χαρτί που λέει απάνω Voting List Heading 5. Τυπωμένο χαρτί μπρος πίσω. Πρώτη τροπολογία. Οριζόντια στρατηγική των εισηγητών για τους μισθούς και τις συντάξεις. Στο παράρτημα Υπάρχουν λεπτομέρειες στον πίνακα 9. Είναι μια οριζόντια τροπολογία η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα εκτός από, τα... εκτός από το Συμβούλιο. Σε όλα τα άλλα θεσμικά όργανα εκτός από το Συμβούλιο. Συμφωνία κυρίων. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια, Standard Abatement Rate. Το ίδιο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια, Έχουμε τις τροπολογίες ε, του εισηγητή για τις άλλες διοικητικές κατηγορίες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται επίση. Οι τρεις αυτές στρατηγικής ε, σημασίας τροπολογίες, οι οριζόντιες, δεν καλύπτουν όμως κάποιες άλλες περιπτώσεις για τις οποίες τώρα θα ψηφίσουμε χωριστά. Πρώτον, 43-96, Ανδρέα Σεν. Κατά εισηγητής, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8805 τώρα, της Γκουε. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κυρία Σούζε, δικιά σας τροπολογία είναι. Δεν είσαστε υπέρ κατά αποχές αποχή κυρία Σούση. Απορρίπτεται λοιπόν. 4577 τώρα. Γρέσλε. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4188 Βέρτμαν. Ο εισηγητη ειναι είναι κατά υπέρ. Κατά, Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία Λίμπε 56-15. Είναι για παρατηρήσεις κατά της διακρίσεων υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε τώρα τρει τροπολογίες τη αναπτυξιακή Επιτροπής. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Ψηφίζουμε μαζί τις τρει τροπολογίες κατά ο εισηγητή. Όχι. Α, όχι λέει η κυρία Σούζα. Ωραία. Πρώτη τροπολογία 5400. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 5406 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5407 υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται επίση. Στη συνέχεια, τροπολογία ΕΛΚ 8262. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεπώς η τροπολογια 4356 καταπίπτει. Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία 82-43. Α, και αυτή καταπίπτει. Σωστά. Οπότε περνάμε τώρα στην τροπολογία της κυρίας Αντρέας. 4409. Ο συγητής είναι κατά, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4410, Ανδρέασεν. Να τις ψηφίσουμε μαζί, 4410 και 4419. Ο συγητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Έχει αποσυρθεί η επόμενη. Και φτάνουμε τώρα στην Ερκιούλ της Γρέσλε. Να μπει σε αποθεματικό. Η Ίγκε θέλει το Hercule 2 να το βάλει και υπέρ στο αποθεματικό κατά. Αποχές μπήκε στο αποθεματικό. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ. Αυτά για την κατηγορία 5 που είναι διοικητικές δαπάνες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τώρα περνάμε στο 3α. Δεν έχω. Bien. Alors. Καλώς. Λοιπόν, εδώ πάρτε το ντοσιέ σας. Αυτό το χοντρό. Στη σελίδα 107 στα γαλλικά τουλάχιστον. Α, όχι, στα αγγλικά. Έτσι καλώς υπάρχει μία. 107 λέει ο πρόεδρος. Σελίδα 107 λοιπόν. 3α. Παρακαλώ. Θέλετε επί της αρχής ψηφοφορία για το να μπει στο αποθεματικό το 75% των γραμμών που έχουν να κάνουν με το Σέγγεν. Έτσι θα κερδίζαμε χρόνο, πιστεύω. Χωρίς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Έτσι, αυτό το είδαμε πριν. Μιλάμε για τις γραμμές που συνδέονται με το Σέγγεν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που το Κοινοβούλιο θέλει να κάνει πάνω σε νέες βάσεις με το Συμβούλιο μετά από το σοβαρό πολιτικό συμβάν που έλαβε χώρα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έθεσε να αμφιβόλο τη συμφωνία που έδωσε στο Κοινοβούλιο το Συμβούλιο Υπουργών για την μεταρρύθμιση του κανονισμού Σέγγεν σε τριμερή διάλογο. Συνεπώς, η διάσκεψη των ε, πρόεδρων των ομάδων μας ζήτησε, και όταν λέω μας ζήτησε, βασικά μας έδωσε την οδηγία, στον προπολογισμό να φανούν οι συνέπειες. Έτσι ώστε να έχουμε ένα μέσο να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο πάνω σε νέες βάσεις υπό τη μορφή μιας πρόταση του να μπει σε αποθεματικό οι σχετικέ γραμμές μέχρι 75%. Σωστά κύριε Σιγητά. Σωστό. Το Συμβούλιο και η Προεδρία θα συνεδριάσουν στις 18 Νοεμβρίου. Και έτσι όπως ζητήθηκε από τους συναδέλφους της ΛΥΜΠΕ, προτείνουμε το αποθεματικό 75% για όλες τις γραμμές, τις τέσσερις γραμμές δηλαδή που εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία. Θέλετε τις γραμμές, να σας τις πω. 297 τροπολογία, 18 0205, 18 είναι τροπολογία 298, Στην 18.05.08 είναι η τροπολογία 308 και στην 18.05.09 είναι η τροπολογία 309. Προ... Προτείνω να ψηφίσουμε ένα μπλοκ. Υπέρ κατά άποχες. Εγκρίνονται αυτές οι τροπολογίες. Τώρα ο εισηγητής θα μου πει αν κάνω λάθος. Αλλά η πρώτη τροπολογία που πρέπει να ψηφίσουμε είναι η 293. Α, ήδη καλύφθηκε. Πάμε στην επόμενη σελίδα. Θα γυρίσουμε σελίδα. Και πάνω στα, στη σελίδα 109 για το σύστημα πληροφοριών Schengen παίρνουμε την τροπολογία 697 της Γκουε που θέλει να καταστραφούν οι γραμμές είναι κατά ο εισηγητής υπέρ. Απορρίπτεται. «318 τροπολογία, χωριστή ψηφοφορία για τα νούμερα και για το ποθεματικό. Είναι υπέρ για τα νούμερα ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατά για το αποθεματικό εισηγητή. Α, είναι υπέρ, υπέρ, υπέρ. Λάθος μου το έπανε, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται επίσης. «7.49 είναι συμβατό». μόνο το αποθεματικό. Αποθεματικό για το 749. Έτσι είναι, κύριε Σιγητά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία 749. Υποθέτω λοιπόν ότι καλύπτει το 43-49. Ωραία. Α, η 800 έχει καταπέσει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Εγκρίθηκε η 297 αποθυματικό Σέγγεν. Ψηφίζουμε για τη 42-25. Συγγνώμη, συγγνώμη. Λάθος. Ψηφίζουμε την 2.97 αλλά μόνο για τα νούμερα γιατί το αποθεματικό το εγκρίναμε. Είναι υπέρο εισηγητής. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για αυτήν τη γραμμή καταπίπτουν οι υπόλοιπες τροπολογίες. 18.02.06 9.78 είναι κατά ο εισηγητής. Ο εισηγητής. για τις 978 και 283 έχουν καλυφθεί. Σε αυτόν τον τομέα πρέπει να ψηφίσουμε μόνο την 298 για τα νούμερα. 298 για τα νούμερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υποθέτω λοιπόν ότι όλες οι υπόλοιπες τροπολογίες της γραμμής ε, καταπίπτουν. Alors, euh, nous passons à European Return Fund. Nous sommes page 111. Σελίδα 111. Τροπολογία ΓΚΟΕ 650. Contre. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Le suivant est identique. Euh, L'amendement 960... 979 ε, των πρασίνων είναι κατά ο εισηγητής. Αποχές, απορρίπτεται. 321 της Λίμπε. Είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 568. Το σύνολο, ε. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 793. Ελκ. Ο εισηγητής είναι κατά. Α, είναι υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ, διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συνεπώς οι δύο άλλες καταπίπτουν. Και έτσι φτάνουμε σε δύο γραμμές που έχουν να κάνουν με τους οργανισμούς και όλα αυτά έχουν ψηφιστεί. Οπότε περνάμε στο Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Τροπολογία 647 της ΚΟΕ. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Αποχές. Απορρίπτεται. 44-55 ήταν ίδια με τα ίδια νούμερα. Απορρίπτεται. 891 των σοσιαλιστών. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά είναι ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. αποχέ Απορρίπτεται. Περνάμε στο επόμενο. Υπάρχουν τρεις ίδιες τροπολογίες. Ο εισηγητής είναι υπέρ. 300 και δύο επόμενες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. σελίδα τώρα 113 στο γαλλικό κείμενο προφανώς. Έκτακτα μέτρα σε περίπτωση μαζική εισρωή προσφύγων. Στα ελληνικά 134. Δύο ίδιε τροπολογίε. 648. Πρώτα η Είναι κατά ο εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτονται. Με συμμαχίε βγαίνει η πλειοψηφία. Τώρα, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών. Τροπολογία 569. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 892 των σοσιαλιστών. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 649 της Γκουέ. Ο συγητής είναι κατά υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Η επόμενη του κύριου Κλήτα είναι η ίδια. Και περνάμε στη 4229. Λάσλο Σουριάν, υπέρ ο συγητής, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και καταβίβει η επόμενη. Στη συνέχεια, όλη η επόμενη σελίδα αντιστοιχεί σε οργανισμούς για τους οποίους ψηφίσαμε ή σε προγράμματα πιλωτικά που θα ψηφίσουμε αύριο. Οπότε γυρνάμε σελίδα και στην ε, επόμενη έχουμε πιλωτικά δοκιμαστικά σχέδια ή οργανισμούς. Οπότε στη σελίδα 117 λέει ο πρόεδρος, στα γαλλικά προφανώς, προετοιμασία... Ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών τη τρομοκρατία. Τροπολογία 741. Σελίδα 140 στα ελληνικά. Κατά ο εισηγητή, ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43-46 του κύριου Άλβαρο. Ο εισηγητής είναι κατά υπέρ. Α, είναι ίδια, είναι ίδια. Συνεπώς απορρίπτεται και αυτή. 308 τώρα. Ψηφίζουμε μόνο τα νούμερα, γιατί το αποθεματικό το ψηφίσαμε ήδη. Ο είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη έχει καλυφθεί έτσι. Επόμενη γραμμή πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας. 284. Κατά ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εδώ πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγώ δεν ψηφίζω λέει ο πρόεδρος. Πέρα στις ψηφοφορίες. 15 υπέρ, 21 ψήφοι κατά, 2 αποχές, απορρίπτεται. 309. Τα νούμερα. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 273 είναι συμβατή, γιατί πρόκειται για θέματα που έχουν να κάνουν με τα δύο φύλλα. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, ο εισηγητής είναι κατά. Ίσως θα πρέπει να μας πείτε το πρώτο τμήμα ποιο ακριβώς είναι και ποιο είναι το δεύτερο, για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Εγώ, λέει ο Πρόεδρος, αντιλαμβάνομαι ότι το πρώτο τμήμα μιλάει εργαλεία για την πρόθεση οριζοντίων μεθόδων και εργαλεία που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο mainstreaming για τα δύο φύλλα και εδώ είναι υπέρ. Α, όχι, κατά διορθώνει ο Πρόεδρος. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου αυτού τμήματος. Κατά. Θα επαληθεύσουμε, νομίζω ότι είναι υπέρ η πλειοψηφία. Ψηφίζουμε, εγώ δεν ψηφίζω. Ψηφίσατε όλοι, ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες. 19 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται. Ε, ενώ είναι ψήφιζα κι εγώ, ε, θα ήταν αποφασιστική σημασία η ψήφος μου. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα τώρα συμπεριλαμβάνοντας λέει, προωθεί πρακτικές για την προστασία των θυμάτων από κλιματικές ενέργειες, ιδίως εκείνοι που έχουν δικές ανάγκες, που είναι θύματα βία σε βάρος των γυναικών, εξαιτία του φίλου κλπ. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Το πρώτο απορρίπτεται, το δεύτερο εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα σε διάφορα δοκιμαστικά σχέδια, το οποίο όμως αφήνουμε για αύριο όπως είπαμε. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών, το κάναμε. Ε, φτάνουμε στο Prince. Είναι προγράμματα που έχουν πολύ ωραίους τίτλους. Ε. Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τώρα, πρίγκιπα Λαβία, Prince Λαβία. 717 προτείνεται να το ψηφίσουμε, αλλά είναι κατά ο Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το ίδιο και το επόμενο. 683 όμως της ΓΚΟΕΣ. Οι είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 310. Υπέρ παρακαλώ. Οι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Επόμενη γραμμή. Αξιολόγηση και εκτίμηση αντικτύπου. 311. Ο συγγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γυρνάμε στη σελίδα. Έχουμε έναν οργανισμό. Προχωράμε. Πάμε στα θεμελιώδη δικαιώματα και ηθαγένεια. Εδώ έχουμε δύο ίδιες τροπολογίες. 894. Ε, κατά ο συγκητής ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 656. Ο συγκητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Με ίδια της κυρίας Βερζιά επόμενη είναι η ίδια, απορρίπτεται και αυτή. 276 τώρα γυναικών. Ο εισηγητής ε, συμφωνεί με τις γυναίκες, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δάφνη τώρα. Έχετε προφορική τροπολογία κύριε Σιγητά για το Δάφνη. Όχι, όχι. Τροπολογία 45-32. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 724 της ΓΚΟΕ. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επίσης με την ίδια πλειοψηφία. 893 τώρα. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται επίσης. 277. Ο εισηγητής είναι κατά υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1016. Ο εισηγητής... Α, είναι ίδια. Είναι ίδια. Άρα πάμε στη 4311 της Βάρμπαρα Ματέρα. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε καλύψει τα επόμενα υπηρεσίες, δηλαδή οργανισμούς ευρωπαϊκούς και δοκιμαστικά σχέδια. Οπότε ερχόμαστε τώρα... Κύριε Σιγητά, ε, δικαιοσύνη, ε. 315, λίμπε. Ο εισηγητής είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Δεν βλέπω χέρια να σηκώνονται, ακούω διάφορα όμως. Κύριε Σιγητά, θέλετε να πείτε κάτι? Στον δικό μου τον κατάλογο είχε συν αλλά τελικά είμαι κατά. Ωραία, 315. Και το μας σημαίνει ότι είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά έχουμε ένα σχέδιο πιλότο. Στη συνέχεια ξαναπάμε στον πρίγκιπα. Είναι η τροπολογία του συγητή. Ο πρόεδρος αποκαλεί τον εισηγητή πρίγκιπα. Είναι η 3311. Και καλύπτει την γραμμή, τη συνέχεια της γραμμής. Πάμε στην 3311 λοιπόν του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται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 Με, ε, ας με παρακολουθεί ο Τζοβάνι, αλλά συμφωνήσαμε χθε με τους συντονιστές για αυτή την κατηγορία 3β να αρχίσουμε ψηφίζοντας την αρχή ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή. Γιατί ζητούμε να ψηφίσουμε αυτή την αρχή. Πρόκειται για μια κατηγορία που έχουμε ελάχιστα περιθώρια για το πλαφόν, για την οροφή και δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ομάδων για την άθρηση των ψήφων. Ξέρετε, η δημοκρατία δημιουργεί αβεβαιότητες πολλές φορές. Εάν τώρα καταλήγαμε εμείς προσθέτοντας τις τροπολογίες να ξεπεράσουμε το πλαφόν, τότε ο εισηγητής θα μας προτείνει να κάνουμε οικονομίες και πιο συγκεκριμένα στο, στα σχέδια πιλότο. Ο καθένας πρέπει να προσέξει να κάνει τους υπολογισμούς του όταν θα πρέπει να Ψηφίσει Ψηφίζουμε λοιπόν να μην ξεπεράσουμε το πλαφόν για το 3β. Ποιος είναι η υπέρ αυτής της αρχής. Je vous remercie. Qui est contre? Personne. Κατά. Αποχές. Η κυρία Σούζα απέχει. Madame Souza aimerait dépasser, mais n'ose pas. <laughs> Bien. Euh, <laughs> ah, Εάν όντως ψηφίσουμε όλε τι τροπολογίε και μετά από του υπολογισμού που θα κάνει η γραμματεία διαπιστώσουμε ότι υπερβαίνουμε την οροφή, τότε θα γίνουν περικοπές στα δοκιμαστικά σχέδια τα οποία θα ψηφιστούν, αλλά όχι στι τροπολογίες. Ναι, ναι, αυτό είναι ο φόβο μου, λέει ο πρόεδρος. Και εγώ το ίδιο αυτό φοβούμαι, λέει ο κ. Γκαριγά. Προχωρούμε τώρα. Με συγχωρείτε, μια στιγμή. Υπάρχει μια τροπολογία πρώτα, υπάρχει μόνο 63 της Επιτροπής Πολιτισμού. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Στο κάτω μέρος της σελίδας είναι δοκιμαστικά σχέδια. Πάλι δοκιμαστικά σχέδια στην επόμενη σελίδα. Προχωρούμε στο πρόγραμμα πολιτισμός. Η τροπολογία 4412, ο εισηγητής αντίθετος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 566, ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 898. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45. Εισηγητής αντίθετος. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 757. Δύο ψηφοφορίες. Πρώτα τα ποσά και μετά το σχόλιο. Ο εισηγητής είναι υπέρ και για τα δύο. Για τους αριθμούς πρώτα, τα ποσά, υπέρ, κατά. Α, αποχές. Εγκρίνονται. Για το σχόλιο, υπέρ, κατά, αποχές. Ίδιο αποτέλεσμα. Εγκρίνεται λοιπόν και αυτό. Και μου λένε ότι το επόμενο έχει καλυφθεί είναι οι γλώσσες που βρίσκονται σε κίνδυνο, άρα δεν είναι πλέον σε κίνδυνο. Προχωρούμε σε προπαρασκευαστική ενέργεια και την ετικέτα ευρωπαϊκής, ευρωπαϊκού πολιτισμού. 66 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Προχωρούμε στα μέσα πέντια κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το 567, ο εισηγητής είναι αντίθετος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το 47 της Επιτροπής Πολιτισμού. Υπάρχουν δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες για τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές. Για τις υποχρεώσεις είναι υπέρ ο εισηγητής, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για τις πληρωμές ο εισηγητής είναι αντίθετος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με πλειοψηφία της δεξιάς και του κέντρου. Ακολουθούν προπαρασκευαστικές ενέργειες και δοκιμαστικά σχέδια και ερχόμαστε στο Media Mundus. 897 εισηγητή υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Είναι κατά ο προσοχή. Κατά. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Ο εισηγητής είναι αντίθετο. Υπέρ. Κατά. αποχέ. ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Η επόμενη ταυτόσημη, άρα απορρίπτεται και αυτή. Άρα, σε αυτή τη γραμμή δεν έχουμε καμία τροπολογία. Απερίφθησαν όλες. Άρα δεν τροποποιείται, δεν τροπολογεί το κοινοβούλιο αυτή τη ε, γραμμή. Για τις ειδικέ αιτήσει εκδηλώσεις, κάτι το οποίο προκαλεί εδώ πολλά πάθη. Έχουμε και έναν πρόσθετο α, πίνακα, τον οποίο ψηφίζουμε όλο μαζί, το Compromise Package. Το έχετε όλοι, γνωρίζετε περί τίνος ψηφίζετε. Ψήφι υπέρ της λίστας των ειδικών αιτήσεων εκδηλώσεων. Κατά. Αποχές. Α, οι πράσινοι απο, απέχουν. Εγκρίνεται ο πίνακας. Αλλάζουμε σελίδα. Νεολαία ενδράση. νεολαία ναι, δράση. Με πληροφορούν ότι ίσως υπάρχει προφορική τροπολογία του εισηγητού. Κύριε εισηγητά. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία να προσθέσουμε ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο ευρώ στις υποχρεώσεις και ένα εκατομμύριο στις πληρωμές. Άρα μιλούμε για τη γραμμή 15-05-55 ένα εκατομμύριο ευρώ και στις υποχρεώσεις και ένα στις ε, πληρώμες. Α, είναι ένα είδος μας, ε, λέει ο πρόεδρος. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα, αυτό καλύπτει όλη τη γραμμή. Έχουμε μετά κάποιες διοικητικές γραμμές και περνούμε στα, στις ενέργειες πολυμέσων. Εδώ η τροπολογία είναι 4181 της κυρίας Βέρτμαν, συγητής αντίθετος, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ο εισηγητής προτιμά την 77 της Επιτροπής Πολιτισμού, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και η επόμενη έχει καλυφθεί πλέον. Ενημέρωση μέσων μαζικής επικοινωνίας. 4182 της κυρίας Βέρτμαν. Ο εισηγητής είναι αντίθετος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ο εισηγητής είναι υπέρ της 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και καλύπτεται και η επόμενη. Για τα κέντρα μετάδοσης πληροφοριών. Εδώ υπάρχει προφορική τροπολογία κύριε Σίγητα. Στην 52 η Επιτροπή Πολιτισμού προτείνει ένα εκατομμύριο υποχρεώσεις, ένα εξακόσα πληρωμές. Εγώ προτείνω να πάμε ένα εκατομμύριο στις πληρωμές. Να βγάλουμε δηλαδή 600.000 από την τροπολογία του, της Επιτροπής Πολιτισμού. Ωραία. Πρώτα να ψηφίσουμε την τροπολογία της κυρίας ε, Βέρτμαν που είναι υπαριθμόν 41-83. Εδώ ο συγητής είναι αντίθετος, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προχωρούμε στην 52 με προφορική τροπολογία του εισηγητού που προτείνει να διατηρηθεί το ποσό στις υποχρεώσεις αλλά να μειωθεί το ποσό των πληρωμών κατά 600.000. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και καλύπτει και την επομένη τροπολογία. Η επόμενη είναι επικοινωνιακή προβολή από τις τη Επιτροπή. 41-84 τη κυρία Βέρτμαν, αντίθετο υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται. 43-16 εισηγητη υπέρ. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Σύμπραξη για επικοινωνιακή προβολή ευρωπαϊκών θεμάτων. 693 της ΓΚΟΕ. Εισηγητής αντίθετος. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41-85. Εισηγητής αντίθετος. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 211 της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων που επιθυμεί βέβαια να προετοιμάσει τις εκλογές αλλά φαίνεται πω όχι ο συγητής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και μάλιστα με ιδιαίτερα υποτιμητικό τρόπο για την ε, Επιτροπή Συνταγματικών. 79 πολιτισμού, εισηγητής υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και καλύπτει, α, πρέπει να ψηφιστούν τα σχόλια ο εισηγητή ε, του ζητού δεν του αρέσουν τα σχόλια. Ψήφι υπέρ των σχολείων. Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Φιλελεύθερη. Ας κάνουμε λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση και εγώ έχω δικαίωμα να ψήφω εδώ, σημειώνει ο πρόεδρος και οι συντονιστές έχουν να πούν τίποτε όχι. Δεν έχει μικρόφωνο ο πρόεδρος, δυστυχώς. Απορρίπτεται τώρα, έχει μικρόφωνο. Ανάλυση και κοινή γνώμη 4186. Ο εισηγητή αντίθετο υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Ο εισηγητή προτιμά την υπαρχόν 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται αυτή και καλύπτει και την επομένη. Προχωρούμε σε επιγραμμικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας. 41-87. Ο εισηγητής αντίθετος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, με τις ίδιες πλειοψηφίες πάντα. 42-53 της κυρίας Πακ. Ο εισηγητής εδώ είναι αντίθετος, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η Ντόρις Πακ θα χαρεί που είδε ότι την ψήφισαν οι σοσιαλιστές. Αυτά τώρα βέβαια ήταν για τα ποσά, για τους αριθμούς. Τώρα είναι ξεχωριστή ψηφοφορία για τα σχόλια. Remarks. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η ομάδα ή μάλλον Ας κάνουμε μια επαλήθευση. Ας κάνουμε επαλήθευση. Άρα, ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα σχόλια. Της 4253. Ο εισηγητής. Ο εισηγητής. Αυτή η τροπολογία είναι ίδια με την 794 ως προς τις παρατηρήσεις. Το σχόλιο είναι το ίδιο. Εγώ ήμουν υπέρ της 794. Δεδομένου ότι ήταν μια τροπολογία που κατέθεσε η ομάδα και όχι μια προσωπική τροπολογία, αλλά μια που λένε τα ίδια πράγματα δεν έχω καμία αντίρρηση. Είμαστε πάντα στα σχόλια της τροπολογίας Doris Pack. Και αν κατάλαβα καλά, ο εισηγητής δε, του δεν του αρέσει η συντάκτρια της τροπολογίας, αλλά δέχεται τα σχόλια. Καλά τα λέω αυτά λίγο για να ασκηθώ. Για να δούμε λοιπόν. Νέα πληροφορία είναι αυτή μπορούμε ίσως να τροποποιήσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Α, α, την διακόπτουμε την προηγούμενη που είχε αρχίσει, διότι δεν είχατε τις σωστές πληροφορίες, φταίω και εγώ ως πρόεδρος. Τώρα είμαστε πια καλά ενημερωμένοι και άρα μπορούμε να ψηφίσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. Μάλιστα, 34 υπέρ 7 κατά θριάμβευσε η κυρία Πακ και ο εισηγητής για τα σχόλια. Τώρα, κατόπιν αυτής, α, ναι, για τα ποσά τώρα πρέπει να ψηφιστεί η 81. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Που έτσι καλύπτει και τις υπόλοιπες. Πάλι μετά ακολουθεί ένα δοκιμαστικό σχέδιο και μετά προχωρούμε στις Ευρώπη, στην Ευρώπη για τους πολίτες. 41-89. Συγητής αντίθετος, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 896. Εισηγητής αντίθετος. Υπέρ. Οι σοσιαλιστές. Κατά. Όλοι οι υπόλοιποι αποχές απορρίπτεται 482 απασχόλησης εισηγητής αντίθετος ψήφι υπέρ κατά απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία όπως πριν ο εισηγητής προτιμά την 82 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προχωρούμε στην επόμενη σελίδα επάνω στην σελίδα, βέβαια στο γαλλικό κείμενο πάντοτε, έχουμε δοκιμαστικά σχέδια και ερχόμαστε στις επισκέψεις στην Επιτροπή. Τι ωραία ιδέα. Έχουμε την υπαριθμόν 83 της Επιτροπής Πολιτισμού για να πάνε να επισκεφθούν την Κομισιόν. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 20 της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών. Υπάρχει προφορική τροπολογία του εισηγητού. 217. Για την 217 αυτή η γραμμή δεν μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Θα μπει στο πακέτο αύριο. Θα ψηφίσουμε τις παρατηρήσεις. Δεν έχουμε ακόμη δηλαδή νομική βάση. Θα ψηφίσουμε δηλαδή για ένα σχέδιο πιλότου ή δοκιμαστικό σχέδιο. Ε, εάν γίνει δοκιμαστικό σχέδιο θα ψηφιστούν τα σχόλια μαζί με το δοκιμαστικό σχέδιο. Αυτό μου φαίνεται λογικό. Άρα προχωρούμε. Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών. Σελίδα 157 στο ελληνικό κείμενο. Το 212. Δεν υπάρχει προφορική τροπολογία. Εάν υπάρχει θα μου πείτε κύριε Σιγητά, έτσι είναι. Πρώτα λοιπόν τα ποσά τα νούμερα δηλαδή και μετά τα σχόλια. Ο εισηγητής είναι κατά των ποσών. Λοιπόν, για τα ποσά, 212 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Για, τα σχόλια, remarks, υπέρ, κατά. Αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για τα σχόλια της 212. Άρχισε η ψηφοφορία. Τώρα τέλειωσε. 19 υπέρ 19 κατά απορρίπτεται. Καλά. Προχωρώ στην 901. Τα ίδια εδώ. Πρώτα τα ποσά, μετά τα σχόλια. Ο εισηγητής είναι αντίθετος. Ποσά, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Σχόλιο, υπέρ, κατά. Ε, υποχρεωτικά θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Ψηφίστε παρακαλώ. Κάθε ψήφος μετρά. Τέλος. Α, 19 υπέρ 20 κατά. Έχει απορριφθεί Τώρα, 400... 290 μάλλον, 290. Ο εισηγητής πάντα αντίθετος. Υπέρ. Α, όχι, είναι, είναι ταυτόσιμη, είναι ταυτόσιμη, με συγχωρείτε. Άρα, 483 Τη επιτροπή Απασχόλησης. Συγητή αντίθετο. Ψήφι υπέρ. Α, άλλαξε γνώμη. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Όχι. Καλά λοιπόν. Είναι υπέρ ο Συγητή. 483. Sorry λέει ο Σύγητης. Τζοβάνι, έχετε το λόγο. Ε, λέει ο εισηγητής, πρέπει να καταλάβετε ότι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Υπάρχει μία προφορική τροπολογία του εισηγητή για την 483 για να προσθέσουμε 500.000 ευρώ για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στις πληρωμές, δηλαδή να πάμε συνολικά σε ένα εκατομμύριο για τις πληρωμές. Η Γιούτα. Γιούτα Χάουκ. Άρα δύο εκατομμύρια στις υποχρώσεις. Α, ένα και ένα. Ένα υποχρώσεις, ένα πλέον. Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, εάν κατάλαβα καλά, τροπολογία 483 επί της οποίας ψηφίζουμε, συνίσταται στα εξής. Ένα εκατομμύριο στις υποχρεώσεις, αυτό δεν αλλάζει, και αντί να βάλουμε 500.000 στις πληρωμές, το κάνουμε ένα εκατομμύριο. Το ίδιο ποσό. Σύμφωνοι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Το επόμενο, η επόμενη τροπολογία καταπίπτει. επικοινωνιακές ενέργειες εν ώψη των ευρωεκλογών, μία νέα τροπολογία της ΑΦΚΟ για μία νέα γραμμή και είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κυρία Σούζα, αποχές, απορρίπτεται. Η υλοποίηση ευρωπαϊκών πρωτοβουλίων πολιτών. Για νέα γραμμή πάλι, είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά έχουμε ένα σχέδιο πιλότο, γυρνάμε σελίδα στο γαλλικό κείμενο. Εδώ έχουμε πάλι δοκιμαστικά σχέδια κλπ. Και πάμε στα Union Action in the Field of Health. 43-34 τα ποσά υπέρ, δεν τα θέλει ο είπε; υπέρ, κατά, αποχέ. απορρίπτεται. Κανεί δεν θέλει τα ποσά. Παρατηρήσει τώρα, remarks. Είναι υπέρ ο συγητής, ποιο είναι υπέρ, κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Επειδή δεν ψηφίζουμε για τα νούμερα, Μπορούμε να ψηφίσουμε την 529 για να αποκαταστήσουμε τα αρχικά ποσά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάλι έχουμε εδώ οργανισμός και έχουμε πάλι πιλωτικά σχέδια, διοικητικές δαπάνες. η Γιούτα λέει ότι ξεχάσαμε μια ψηφοφορία. No. Ε, Όχι. Αν συμφωνεί ο εισηγητής, πάμε στη σελίδα του γαλλικού κείμενου 135, 134, πολιτική προστασία της, εντός της Ένωσης Έχουμε μία τροπολογία του Γιώργου Σταυρακάκη και είναι υπέρο Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τελειώσαμε με το 3β. Θα κάνουμε τώρα την πρόσθεση για να δούμε αν είμαστε στα όρια της οροφής και προτείνω δύο λεπτά για να προετοιμάσουμε την ψηφοφορία για την κατηγορία 2. Bien. Everybody has had Λοιπόν, εντάξει, όλοι πήρατε μια ανάσα. Μπορούμε να αρχίσουμε και πάλι. Κατηγορία 2. Σελίδα 80, στο γαλλικό προφανώς αντικείμενο. Συνεπώς, μέχρι να επιστρέψει το ΕΛΚ. Ναι, έχουν πάει να πλύνουν τα χέρια τους, ναι. Λέει ο Πρόεδρος. Για μια συμφωνία με τον εισηγητή. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, που είναι αρκετά γρήγορος και για την κατηγορία 2, και αν στο μεταξύ έχουμε τυπώσει όλες ε, τις ψηφοφορίες για την κατηγορία 4. Θα μπορέσουμε σήμερα να ψηφίσουμε και για την 4. Σας το λέω ώστε οι συνεργάτες μας να ξέρουν ότι μπορούν να πάνε και να τυπώσουν τους καταλόγους ψηφοφορίας και για την κατηγορία 4. Συμφωνεί. Κατηγορία 2 τώρα. Ησυχία παρακαλώ. Λοιπόν, κατηγορία 2. Κύριε Σιγητά, μπορούμε να ψηφίσουμε γραμμή-γραμμή ή θέλετε να μας προτείνετε πρώτα κάτι, μια προφορική τροπολογία ή κάτι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, όπως γνωρίζουν και οι συντονιστές, πολλές φορές είχαμε την ευκαιρία μέχρι τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που έχει να κάνει μετά τα αποθεματικά. Και για πρώτη φορά στην κατηγορία 2 θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για τις γραμμές που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Το ίδιο πρόβλημα όμως θα τεθεί και αύριο όταν ψηφίσουμε την 1β. Έχουμε επιφυλάξεις που έχουν υποβάλει οι σοσιαλιστές αλλά και οι φιλελεύθεροι. Από τους σοσιαλιστές μου ζητήθηκε να αναλάβω εγώ και να παρουσιάσω προφορική τροπολογία. Πρέπει να κάνουμε διάφορες γραμμές 04, 02, 06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 100% στο αποθεματικό των πιστώσεων πληρωμών για κάθε γραμμή. Και για προϋπόθεση η κυρία Γαρδία Μπαζάλ, προκειμένου δηλαδή να απελευθερωθεί το αποθεματικό αυτό, εκείνη θα μας ενημερώσει. Γιατί εκείνη έχει δουλέψει πάνω σε αυτό πιο πολύ. Ωραία, έχετε πάρει όλοι το χαρτί, έτσι. Έχει μοιραστεί. Εδώ είναι όλες οι γραμμές οι οποίες έχουν να κάνουν με τα αποθεματικά αυτά. Αυτά που μόλις μας διάβασε ο εισηγητής και που αναφέρουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αρθεί το αποθεματικό. Μπορείς να μας παρουσιάσεις, παρακαλώ. Ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις. Το το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και οι συντονιστές και στην Επιτροπή. Πάντως στόχος του αποθεματικού αυτού είναι να πετύχουμε ενημέρωση από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή βέβαια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τις πληρωμές. Επίσης δεν θέλουμε ποτέ να φτάσουμε με το αποθεματικό αυτό στην ε, συνδιαλογή. Θέλουμε μια θετική ανταπόκριση από το Συμβούλιο ώστε να ζητήσει από το Κοινοβούλιο να αυξηθούν οι πληρωμές για το 2013. Καλώς, Σαλβαδόρ. Ναι, το συζητήσαμε οι συντονιστές. Το κατά πόσο πρέπει όχι να υπάρξει αυτό το παθηματικό. Η πολιτική μου ομάδα εξακολουθεί να είναι κατά κάποιου τέτοιου είδους αποθεματικού ή δέσμευση τέλο πάντων των δαπανών όσον αφορά την συνοχή και τα διαφορετικά ταμεία. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτό προσφέρει κάτι και εξάλλου θα είναι δύσκολο να εξηγήσουμε ότι για να σώσουμε τις πληρωμές τελικά χρησιμοποιούμε χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία. Η ομάδα μου λοιπόν δεν συμφωνεί, αλλά συμφωνούμε να ψηφιστεί. Είναι μια προφορική τροπολογία, δεν έχουμε αντίρρηση, να τεθεί σε ψηφοφορία εφόσον την υπογράφουν δύο σημαντικές μεγάλες ομάδες. Οπότε να ψηφίσουμε. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Αυτή είναι μια υπόθεση που έχουμε συζητήσει πράγματι επί μακρός τους συντονιστές. Είναι ένας τρόπος να δούμε κάπως διαφορετικά το θέμα και το πρόβλημα των ε, πληρωμών. Επιπλέον, πρέπει να σας πω, είμαστε σε μια συνεδρίαση που πώς γνωρίζετε, ε, περνάει και μεταδίδεται και στο διαδίκτυο, έτσι. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι την πρωτοβουλία μας είχαμε μια τριμερή συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο καταρχήν και μετά και σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στην Προεδρία του Συμβουλίου, τον Κυπριπουργό, τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι και την Επιτροπή Προπολογισμών. Όλες οι ομάδες ήταν παρούσες με κάποιον εκπρόσωπο. Και αυτό για να διευκρινίσουμε τον τρόπο υπολογισμού των αναγκών σε πληρωμές έτσι όπως το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των ποσών που στέλνουν τα κράτη-μέλη. Μας επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι ο καθορισμός αυτός των ποσών των αναγκών σε πληρωμές γίνεται μέσα σε μεγάλη σύγχυση και χωρίς καμία διαφάνεια, ούτε σαφήνεια. Και όπως το είπα και χτες στους συντονιστές, έδωσε μια συνέντευξη τύπου ακριβώς για να δώσω μια περίληψη στον τύπο των συμπερασμάτων στα οποία είχαμε καταλήξει μετά από αυτήν την τριμερή συνάντηση και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από διάφορες χώρες που ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό αυτό ε, θα βοηθήσουν στο να γίνουν διαφορετικά από ό,τι έγιναν πέρυσι γιατί πέρυσι είχαμε παραμείνει σε μια πλήρη σύγχυση όσον αφορά τις πληρωμές μέχρι την τελευταία στιγμή των διαπραγματεύσεων. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι απαράδεκτο πολιτικά. Αυτή είναι μια περίπλοκη βέβαια διάσταση. Δίχως άλλο πάντως, θα μας οδηγήσει στο να εισαγάγουμε τρόπο ίσως στο δημοσιονομικό κανονισμό. Αν μη τι άλλο, στα πλαίσια του πολιετούς ε, πλαισίου και στην διοργανική συμφωνία. Γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να έχουμε έναν τέτοιο διάλογο κοφών όσον αφορά τις πληρωμές και εμείς, Κοινοβούλιο, να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εντελώ παράλογη γιατί αναγκαζόμαστε να στηρίξουμε επιστώσεις πληρωμών που δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες του Κοινοβουλίου, στα χρήματα του Κοινοβουλίου, στην πολιτική του Κοινοβουλίου, αλλά σε επιστροφές, αποζημιώσεις που χρειάζονται τα ίδια τα κράτη-μέλη. Είναι μια κατάσταση παράλογη. Αυτά. Από εκεί και πέρα. Ο εισηγητής, από ό,τι καταλαβαίνω, μας υποβάλλει μια προφορική τροπολογία, που δεν υποστηρίζει όμως ο ίδιος, ε? δεν την υποστηρίζει. Αλλά που λέει ότι πρέπει να ψηφιστεί. Να την ψηφίσουμε. Παρακαλώ κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εκφράσατε σαφέστατα τη θέση μου. Εγώ είμαι υπέρ της ψηφοφορίας, της προφορικής τροπολογίας, η προσωπική μου γνώμη είναι αντίθετη. Αυτή η τροπολογία αντικαθιστά αυτήν την οποία ψηφίζουμε και τις άλλες τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί για το αποθεματικό και για τις οποίες πρέπει να ψηφίσουμε αύριο. Δεν θα ήθελα να ψηφίζουμε πολλές φορές παρόμοια πράγματα. Με άλλα λόγια, θα ψηφίσουμε σε αυτές τις γραμμές για τα νούμερα. προτείνονται τροπολογίες για να μπει στο αποθεματικό το σύνολο των πιστώσεων ορισμένων γραμμών. Εάν εγκριθεί η τροπολογία, δεν θα ψηφίσουμε πια για τα αποθεματικά αυτών των γραμμών. Είναι φανερό. Όλα μπαίνουν στο αποθεματικό. Αλλά μπορούμε να έχουμε γραμμές για τις οποίες αν έχει αν απορριφθεί η τροπολογία και έχουμε μια πρόταση να μπει το 20% στο αποθεματικό, τότε θα πρέπει να ψηφίσουμε. Ή δεν θα συμβεί αυτό. Σύμφωνοι? Ε, Ιντερ, έτσι καταλαβαίνετε, κατανοείτε τα πράγματα βέβαια. Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση, διότι αυτές οι προφορικές ε, τροπολογίες αντικαθιστούν τις τροπολογίες που είχαμε καταθέσει, αλλάζουν τα σχόλια, εμείς ζητούσαμε 100% στο ποθηματικό. Θα ήταν βλακεία να τις ψηφίσουμε και πάλι. Δεν έχει νόημα. Ωραία. Αυτό απλουστεύει τα πράγματα. Αποσύρετε εσείς τις τροπολογίες για τα αποθεματικά ε, ε, και έχουμε αυτή την προφορική τροπολογία ή όλα ή τίποτα. Ο εισηγητής για τους σοσιαλιστές είναι σαφής η διευκρίνηση ότι ε, αυτή η προφορική τροπολογία αντικαθιστά και καταπίπτουν όλες οι άλλες. Αλλά ρωτώ τους φιλελευθέρους, το ίδιο ισχύει και για τη δική τους τροπολογία που κατέθεσαν για το αποθυματικό. Ποιος θα μιλήσει για τους φιλελεύθερους, γιατί δύο ζήτησαν το λόγο. Ο Γιάν Μούλτερ. Ο Γιάν. Όσον αφορά τους φιλελεύθερους, όσον αφορά τους φιλελεύθερους, εμείς θα υπερψηφίσουμε. Θέλουμε να ψηφιστεί η τροπολογία, θα την υπερψηφίσουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι ισχύει το ίδιο και για τα άλλα. Ε, that means that we keep as liberals our εμείς διατηρούμε την τροπολογία που προτείναμε για το αποθεματικό, εμείς ως φιλελεύθεροι. Καλώς, Έλγα και μετά εισηγητής, Έλγα, για την πολιτική προσέγγιση της δικιάς μου ομάδας. Βεβαίω για μένα είναι εντάξει να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία, δεν τίθεται θέμα, αλλά όπως έχω ήδη πει, εδώ δίνουμε αγώνα για το επίπεδο των πληρωμών. Και αυτή η προφορική τροπολογία για 100% στο αποθεματικό για μένα είναι πολύ δύσκολο να το περάσουμε στον έξω κόσμο. Δεν είναι το σωστό μήνυμα δηλαδή που θα στείλουμε στον κόσμο και γι' αυτό και θα την καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ξεκάθαρο. Ο εισηγητής. Εγώ ε, θέλησα το λόγο γιατί επειδή έσβησε το μικρόφωνο του κύριου Μούλτερ δεν είχα καταλάβει τι θέλαν να κάνουν οι φιλελεύθεροι με το απόθεμα. Οπότε είναι πλέον σαφές ότι θα ψηφίσουμε. Οι σοσιαλιστές αποσύρουν την τροπολογία που θα ψηφίζαμε για το 1β αύριο το πρωί, γιατί αφορά στο ίδιο αποθεματικό, ενώ οι φιλελεύθεροι προτίθενται να διατηρήσουν την τροπολογία τους. Θα την ψηφίσουμε όμως αύριο όταν έρθει η ώρα. Πολύ ωραία. Εφτά προφορικές τροπολογίες που έχουν καταθέσει δύο ομάδες. Θέλει να τις ψηφίσουμε ο εισηγητής υπέρ, αλλά δεν τις υποστηρίζει. Μπορώ να ψηφίσω. Όχι, υπάρχει άλλος. Δεν μπορώ. Ωραία. Δεν μετράει ψήφο. Μου είπαν όχι, έχει δύο πεπέ παραπάνω. Ωραία, αρχίζει η ψηφοφορία και δεν ψηφίζω. Και άλλος ε, Πέπε, άλλος του ΕΛΚ είναι παραπανήσιος. Παρακαλώ κάποιον να μην ψηφίσει. Η κυρία Καρβάλιο λοιπόν απέσυρε. Όλοι οι παρόντες ΕΛΚ μπορούν να ψηφίσουν πλην της κυρίας Καρβάλιο και του Προέδρου. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Δεν υποχρεούνται, αλλά έχουν δικαίωμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. 17 υπέρ 23 κατά και δύο αποχές. Δεν εγκρίνεται η προφορική τροπολογία. Απέσυρε η σοσιαλιστική ομάδα τη δική της τροπολογία, οι φιλελεύθεροι διατηρούν τη δική τους. Πάμε τώρα. Στην κατηγορία 2, σελίδα 91 στο γαλλικό κείμενο, ξεκινάμε με ένα δοκιμαστικό σχέδιο και πάμε στην τροπολογία 998 και είναι κατά ο εισηγητής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 685 42-41 είναι ίδιες απορρίπτονται 34 της Γεωργίας υπέρ ηγητής κατά έχει γνώμη το ΕΛΚ Είναι υπέρο εισηγητής. Κατά. Τροπολογία 34. Ναι, είναι για τους ε, αγρότες, ξέρετε. Αποχές. Εγκρίνεται με συγκεχημένο τρόπο. «591 Programs for Private Persons» υπερκατά αποχές απορρίπτεται 999 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42-30 είναι κατά ο εισηγητής υπέρ κατά αποχές ε, ε θα ελέγξουμε Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 15-24 απορρίπτεται. Όλες οι τροπολογίες για αυτό το πρόγραμμα απορρίπτονται. Ζάχαρο και ιζογλυκόζι. Ο Ντέρεκ θέλει να πει κάτι. Εγώ έχω έξι πολύ παρόμοιε τροπολογίες για επιστροφές εξαγωγών. Ας κάνουμε μία ψηφοφορία για όλες μαζί. Αυτήν την τροπολογία και τις ε, ίδιες τροπολογίες του Ντέρεκ. Υπέρ. Είναι κατά ο εισηγητής. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με σκλη... στεναρή πλειοψηφία. Ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών για προ... προαναγνώριση. 18 είναι υπερουσυγητής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλύπτονται όλες οι υπόλοιπες. Επόμενη σελίδα. Σχέδιο πρόθεσης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία 16 της ΓΚΟΕ κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτει και το επόμενο. 19 της Άγκρη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν όλες οι υπόλοιπες τροπολογίες. Αμπελοϊνικό τομέας. Επιτέλους κάτι το ενδιαφέρον, λέει ο πρόεδρος. 4108. Είναι κατά ο εισηγητής. Έκπληξη. Υπέρ. Κατά. Όσοι αγαπούν το κρέας είναι κατά. Αποχές απορριπτεται 4151 είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Τρεις. Οι βόρειοι και οι νησιώτες κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στα λοιπά μέτρα. 41-07. Κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 41-52 υπέρ. Η συνήθιση ύποπτη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απόλυτα λογική ψηφοφορία. Ενέργειες προώθησης, πληρωμές από τα κράτη-μέλη, 20. Είναι κατά ο εισηγητής. Α, είναι υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ, κατά ποχές εγκρίνεται. Καλύπτει όλη τη γραμμή. Πάμε στις αποξηραμένες ζωοτροφές. 41-53 είναι κατά ο εισηγητής. Κατά, απορρίπτεται. Γάλα και γαλακτοκομικά. 31 της Άγκρη, τον υποστηρίζει ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καρύπτει όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες. Γάλα για τους μαθητές. 876 είναι κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4178 η Υγεία. 617 της ΓΟΥΕ, Είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Ηλεκτρονικά. Διότι εδώ ξεπερνάει τα όρια της κλασικής αριστεράς. Μπορώ να ψηφίσω ρωτάει ο πρόεδρος. Ναι. Πολύ μυστηριώδες όλο αυτό. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ 24 κατά. Είμαι υπέρ του school wine, κρασί στα σχολεία και όχι γάλα λέει ο πρόεδρος. Και η πολιτική μου καριέρα θα σταματήσει εδώ. Απορρίπτεται. Κλούτε είναι η ίδια, 42-31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Βόλιο κρέας. 9-98, ε, είναι κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 33 της Άγκρη είναι υπέρ εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γυρνάμε σελίδα. Ζώντα ζώα. Αυτό με ενδιαφέρει, έχει πλάκα, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, έχουμε ενισχύσεις και για τα πεθαμένα ζώα και για τα ζωντανά ζώα. Για τις αμβλώσεις τα ζώα δεν έχει ενίσχυση, για τα ζώα που θα γεννηθούν ούτε. 32. Την υποστηρίζει ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όλες οι υπόλοιπες καταπίπτουν. Για τα γουρούνια τώρα, λέει. Είναι, είναι υπέρ των γουρούνιων, υπέρ των χείρων ο εισηγητής. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τα γουρούνια στο 30, λέει ο πρόεδρος. Πάμε στα αυγά, ο μελέτες. 39 που είναι υπέρ ο εισηγητής. Ποιος είναι υπέρ της ομελέτας. Κατά. Κανένας. Όλοι αγαπούν τα αυγά. Ομόφωνα περνάει η 39. Πάμε στα κοτόπουλα. Κρέας πουλερικών. 998 είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Λάθος έκανε. απορρίπτεται. Καλύπτονται και οι υπόλοιπε τροπολογίε. Πάμε στην 29 της Άγκρη. Είναι υπέρ ο εισηγητή. Υπέρ. Το ΕΛΚ μπορεί από καιρού ει καιρό να σηκώνει το χέρι του. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Μέλισσες ειδικε ενισχυσει ενισχύσεις. 41-56 είναι κατά ο εισηγητή. Υπέρ. Κατά των μελισσών. Σα ευχαριστώ. Αποχέ. απορρίπτεται. <laughs> Από μία πλειοψηφία ασιατικών κυφήνων, λέει ο Πρόεδρο. Συριαν υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, τα, τα, λίγο διότι οι ομάδες έχουν διασπαστεί για τις μέλισσες αλλά υπάρχει μια πλειοψηφία κατά. Η θνησιμότητα των μελισσών θα συνεχιστεί. Λοιπόν, μετά έχουμε δοκιμαστικά σχέδια και πάμε εδώ. Έχουμε μία ένα... Α, ξαναπάμε στα βοηδή. Ειδική πρημοδότηση για βοηδή. Για τα bullfighting εδώ. Έχουμε ταυρομαχίες ε, υπέρ. Ιαν. Θα σας πω το ίδιο που είπα και πέρυσι. Αυτό το ποσό δίνεται στη Δανία, στη Σουηδία και νομίζω τη Σλοβανία ή την Σλοβακία. Δεν νομίζω ότι έχουν τα δρομαχίες εκεί. Όχι, απλώς για να εξηγήσω το πόσο εμείς θα ψηφίσουμε. Και ψηφίζετε δηλαδή υπέρ ή κατά. Κατά. Καλώς. Έλεγα. Ναι, αλλά εδώ λέω ότι τα χρήματα δεν πρέπει να πάνε σε ταυρομαχίες, οπότε εντάξει για μένα. θανατηφόρες. Α, γιατί υπάρχουν χώρες όπου παίζουν, δηλαδή έχουν ένα παιχνίδι, δεν τους σκοτώνουν τελικά τους τάβρους. Α, μην γελάτε, ναι, έτσι είναι. Να, στην Πορτογαλία για παράδειγμα γίνεται κάποιο είδος σταυρομαχίες όπου δεν θανατώνεται ο τάβρος. Πρέπει εδώ να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, έτσι. Δεν είναι για γυαλιά. Για μερικούς από εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία για αυτή την τροπολογία. Και εδώ επιμένει ιδιαίτερα ο συντονιστής μας του ΕΛΚ. Ψηφίστε, ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. 13, υπέρ της τροπολογίας, 27 κατά. Απορρίπτεται. Καπνός. Όλα τα προβλήματα τάβρων, ε, βοδιών και αγελάδων τα λύσαμε. Και τώρα πάμε στο τοπάρισμα λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, υπέρ της πρώτης τροπολογίας. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Καπνίζει, καπνίζει, καπνίζει και ο καπνός είναι μαύρος. Απορρίπτεται. 21 ε, κατά 17 υπέρ. Δεν θα έχουμε λοιπόν τροπολογίες για τον καπνό. Ειδική στήριξη. Συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. Πρόκειται για τη βοήθεια στα ζευγάρια, ενισχύσει στα ζευγάρια ή για τις ζευγμένες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γυρνάμε σελίδα 90 στο γαλλικό κείμενο προπαρασκευαστική ενέργεια, θα το δούμε αύριο. Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, 618 της ΓΚΟΥ είναι κατά ο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφτεται. 4484. Το ίδιο. 910. καλύφθηκε, έχει ψηφιστεί. Οι σοσιαλιστές τα πέσυραν. 24 100 εκατομμύρια. Είναι υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπάρχει ένα σχόλιο για το 10.02. Ε, Πρέπει να ψηφίσουμε το σχόλιο και ο εισηγητής είναι κατά. Για το σχόλιο του 10.02 η Έλγα είναι υπέρ. Κατά. Πολύ. Αποχές. Απορρίπτεται το σχόλιο. Μετά έχουμε ένα δοκιμαστικό σχέδιο. Λογιστική εκαθάριση. 509. Της Επιτροπής Περιβάλλοντος και είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται και άλλες δυο. 25 της Άγρη είναι υπέρ ο εισηγητής υπέρ. Κατά αποχές, πλειοψηφία υπέρ, εγκρίνεται. Επίλυση διαφορών, τροπολογία της κυρίας Ανδρεάσιν, είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινή γεωργικής πολιτικής, ευγενές σχέδιο. 576 είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 22, υπέρ είναι υπέρ ο εισηγητής. Κατά. Απορρίφθηκε, αλλά να το επαληθεύσουμε. Ψηφίζω κι εγώ. Ψηφίστε. Πέντε κοιμούνται, λέει ο πρόεδρος. Πέρας ψηφοφορίας. πέντε υπέρ 21 κατά απορρίπτεται η τροπολογία. Ψηφίζουμε την 510 Είστε υπέρ ή κατά εισηγητά. Είναι υπέρ. Ναι, ναι. Υπέρ της 510. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλύπτει και την επόμενη τροπολογία αυτή. Αφήνουμε, στο δοκιμα... Αφήνουμε το δοκιμαστικό σχέδιο και πάμε στο Life Plus. 587 είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 710 της ΓΟΥΕ. Κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 624 της ΓΟΥΕ είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές ίδιος συσχετισμός για πόρυψη. Ο εισηγητής προτιμάει την 535 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καλύπτονται όλες οι υπόλοιπες. Λοιπόν, έχουμε δοκιμαστικό σχέδιο και ευρωπαϊκούς οργανισμούς δοκιμαστικός ευρωπαϊκός οργανισμός πάλι έχουμε εδώ δοκιμαστικά σχέδια και οργανισμούς και πάμε στις παρεμβάσεις για τα προϊόντα αλίας διότι όλα τα υπόλοιπα έχουν καλυφθεί από την προηγούμενη ψηφοφορία 708 της Γκουε είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται, έχει απομονωθεί η Γκουε. 4504 είναι ίδια. Σχέδιο ε, δοκιμαστικό σχέδιο, πρόγραμμα αλίας για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. 713 Είμαστε για τις απομακρυσμένες περιφέρειες, τα ΙΤ, η νησιά του Ειρηνικού, η προτείνει την 713 κατά εισηγητής υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και η επόμενη επίσης. Πάλι έχουμε δοκιμαστικά σχέδια, όλη η σελίδα είναι δοκιμαστικό σχέδιο. Και πάμε στις προπαρασκευαστικές εργασίες των νέων διεθνών οργανισμών αλληλείας κλπ. 3.27. Είναι κατά ο εισηγητής. Ψήφι υπέρ. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά διότι δεν σηκώνονται πολλά χέρια. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ένα σοσιαλιστής παραπάνω. Μία ψήφο σοσιαλιστών παραπάνω. Η κυρία Τρότμαν βγάζει την κάρτα της. Εντάξει. Καλά λοιπόν, τέλειωσε η ψηφοφορία και το αποτέλεσμα είναι 14 υπέρ 24 κατά. Έχει λοιπόν απορριφθεί. Ενίσχυση διαλόγου με βιομηχανία αδείας εννοείται. 228 εισηγητής είναι αντίθετο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλλήλεια 707. Εισηγητής αντίθετος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και συμπαρασύρει και την επόμενη που είναι ε, ισοδύναμη. Τώρα, Σελίδα 100 στα γαλλικά, 120, 120 στα, στο ελληνικό κείμενο. 628 της ε, Ενωτικής Αριστεράς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44-74 Α, το ίδιο, είναι, πρόκειται για το ίδιο κείμενο 911 απόσυρση του αποθεματικού Άρα προχωρούμε στην 329 Επιτροπή Αλληλεία. Συγητή είναι σύμφωνο ή ψήφι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Και καλύπτει και την επόμενη. Εκτός στόχου σύγκριση τώρα. Υπάρχουν λοιπόν οι στόχοι σύγκριση και εκτός στόχων σύγκριση. 629. Ο Συγητή αντίθετος. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη ήταν α, ταυτόσημη. Η 912 ήταν αποθεματικό σοσιαλιστικό το οποίο έχει εξαφανιστεί τώρα και ψηφίζουμε λοιπόν την 330 ο εισηγητής είναι σύμφωνος, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά ακολουθούν ορισμένα δοκιμαστικά σχέδια και ερχόμαστε στην στήριξη για τη διαχείριση ελευτικών πόρων. Τροπολογία 577 των ε, συντηρητικών. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 679 ενωτικής αριστεράς. Συζητής αντίθετος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4506 ταυτόσημη. 331 Επιτροπής Αλίας εισηγητής αντίθετος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Πρόκειται για διάσπαση των ομάδων. Ας κάνουμε μια επαλήθευση. Μια στιγμή, μια στιγμή δεν βλέπω. Υπάρχουν παραπάνω σοσιαλιστικές ψήφοι. Όχι, μπορείτε να ψηφίσετε όσοι θέλετε. Καλά. Πέρα τη ψηφοφορία τώρα και το αποτέλεσμα είναι 15 υπέρ, 24 κατά. Άρα απορρίπτεται. Απορρίπτεται όπως είπα. Άρα για τη γραμμή αυτή δεν υπάρχουν τροπολογίες. Και ακολουθούν ορισμένα δοκιμαστικά σχέδια και ερχόμαστε στην 332. Εισηγητής αντίθετος, ψήφι υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση. Τα χέρια δεν σηκώνονται πια αρκετά. Πέρας. 13 υπέρ 26 κατά, άρα απορρίπτεται. Και ακολουθεί, ακολουθούν ορισμένες, ορισμένοι οργανισμοί και ακολουθεί πρόγραμμα με στόχο τη στήριξη περαιτέρω ανάπτυξη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. 335 Επιτροπή Αλληλεία. Εισηγητή είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Άρα καταπίπτουν οι υπόλοιπε. Ακολουθούν δοκιμαστικά σχέδια. Νέα μέτρα για φυτοϊγειονομικές παρεμβάσεις. 709 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 518. Εδώ προτείνεται ...709. Θέλετε ψηφοφορία κατά τμήματα για τα σχόλια του 709. Ο εισηγητής τι νομίζει, ο εισηγητής... Και σε αυτή την περίπτωση η 709, 518 όπως και οι 4505 έχουν τις ίδιες παρατηρήσεις. Η θέση του εισηγητή είναι αρνητική για τα ποσά, αλλά είμαι υπέρ των παρατηρήσεων. Καλά λοιπόν. Σχόλια. 709. Ο συγητής είναι σύμφωνος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για την 518. Εδώ πρέπει να ψηφιστούν τα ποσά. Όχι. Α, ε, καταπίπτει αυτή. Καταψηφίστηκαν τα ποσά της 709. Και εδώ οι αριθμοί, τα νούμερα είναι διαφορετικά. Άρα νομίζω δεν ψηφίσαμε προηγουμένως τα ποσά, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε, πρέπει να ψηφίσουμε τώρα τα ποσά. Είτε υπέρ είτε κατά, αλλά πρέπει να συζητηθούν. Συμφωνείτε καλά λοιπόν, ωραία. Για τα ποσά λοιπόν τώρα, 518. Εισηγητή αντίθετο ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Προχωρούμε τότε στην 27. Εισηγητή αντίθετο. Α, υπέρ. Είναι υπέρ. Καλά. Είναι υπέρ ο εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Και καλύπτει τα υπόλοιπα. Τι υπόλοιπε τροπολογίε. Και έχει τελειώσει εδώ η κατηγορία 2. Διακοπή λοιπόν. Κύριε Σιγητά, εσείς πρώτα. Νομίζω ότι οι ομάδες δεν έχουν ετοιμάσει ακόμη τον κατάλογο ψηφοφορίας ε, για, την, ε, για, ε, για, τον τομέα 4, οπότε θα πρέπει ίσως να τον αναβάλουμε για αύριο το πρωί. Τι λένε οι ομάδες. Οι σοσιαλιστές είναι, οι σοσιαλιστές είναι έτοιμοι. Οι φιλελεύθεροι είναι έτοιμοι. Έτοιμοι. Οι πράσινοι είναι έτοιμοι. Οι ECR είναι έτοιμοι. Και η Μάρτα Ανδρέας είναι έτοιμη επίσης, ίσως όχι να υπερψηφίσει, αλλά έτοιμη να ψηφίσει. Μόνο το ΕΛΚ δεν είναι έτοιμο. Κυρία Σούζα, είστε έτοιμοι. Ε, we are not ready as... Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, αλλά πολύ σύντομα θα είμαστε. Πρόεδρος, ωραία, να διακόψουμε για πέντε λεπτά να ελέγξουμε, να βεβαιωθούμε ότι είναι όλοι έτοιμοι και η δικιά μου η ομάδα. Έτσι σε πέντε λεπτά. Okay. Ladies and gentlemen. Καλώς, λοιπόν. Ελέγξαμε και είδαμε ότι όλες οι ομάδες είναι έτοιμες τώρα. Υπάρχουν οι κατάλογοι ψηφοφοριών λοιπόν για όλες τις πολιτικές ομάδες. Όλοι εκτός από μένα. Εγώ δεν είμαι έτοιμος, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίας λοιπόν. Και αρχίζουμε με ψηφοφορία συνολικά κάποιου συμβιβασμού, ε, του συμβιβασμού. Συμβιβασμός ο οποίος έχει να κάνει με τα ποσά μόνο. Υπάρχουν λοιπόν τρία κομμάτια. Πρώτο υποτμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. First subblock. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο subblock. Για επιστροφή του σχεδίου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τρίτο οι split lines, χωριστές γραμμές. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνεπώς, οι ψηφοφορίες αυτές που κάναμε για όλα μαζί περνάνε. Τώρα περνάμε στις χωριστές ψηφοφορίες που δεν καλύπτονται από το συμβιβασμό και πάντα μόνο τα ποσά 01, 03, 2 γραμμή. Τροπολογία 41-40. Ο συγητης ειναι είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89-22 κατά εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. 88-29 της ΚΟΕ. Διαφωνεί ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88-11. Και άλλες δύο που είναι ίδιες. Ε, πάλι διαφωνεί ο εισηγητής υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88-12. Ο εισηγητής διαφωνεί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με ίδιες πλειοψηφίες. 88-33 διαφωνεί ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88-01. Ο εισηγητής διαφωνεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85-52. Διαφωνεί ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε τώρα στην 8802 της ΓΚΟΕ εναντίον εισηγητής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8094. Δεν ψηφίζουμε παρά μόνο τις πληρωμές για να επαναφέρουμε το σχέδιο προπολογισμού. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στα σχόλια. 42-38. Ανταλλαγέ εμπειρογνώμων. Υπέρ ο Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζω, έτσι, εκτός αν μου το απαγορεύσουν. Δεν είναι εδώ κυρία Τρότμαν. Μπορούν ε, οι σοσιαλιστές να ψηφίσουν άνετα, λέει ο πρόεδρος. Πέρας της ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται η τροπολογία. Ερχόμαστε τώρα στην 86-72. Ο εισηγητής διαφωνεί. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. 87-85 τώρα. Εδώ κατά τμήματα ψηφίζουμε. Πρώτο τμήμα. Whole new text. Νέο κείμενο που έχετε. Ο συγκτής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Έχει νόημα, αν λείπει το πρώτο τμήμα, να ψηφίσουμε το δεύτερο. Όχι, έτσι. Όχι, δεν έχει νόημα. Συνεπώ, χωρί πρώτο τμήμα δεν υπάρχει ούτε και δεύτερο. Ακέφαλο ψάρι δεν μπορούμε να έχουμε. Συμφωνούμε, έτσι. Ωραία. Πάνω όλα αυτά. Συνεπώ, περνάμε στην τροπολογία τη ΑΦΕΤ, εξωτερικών υποθέσεων, 51-66. Για να αλλάξουμε τον τίτλο της γραμμής. Υπέρ, συμφωνεί και ο συγκριτής. Κατά, αποχές, Απορρίπτω. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Γκουε 8801. Όχι χρηματοδότηση για δράσεις στρατιωτικού χαρακτήρα. Υπέρ παρακαλώ, ο Σύγκριτης διαφωνεί. Της Γκουε. Κατά. Απορρίπτεται. Γυναικών 6207. Ο εισηγητή διαφωνεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4274. Για την πρόθεση της μη βίας. Ο εισηγητής διαφωνεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 86-73 πρασίνων. Ο εισηγητής διαφωνεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία ΕΛΚ 82-17. Συνδυτοποίηση κατά προτεραιότητα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο εισηγητής συμφωνεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα του εισηγητή. Την δημιουργία ενός δικτύου και διευκόλυνσης για διαμεσολάβηση και διάλογο και ε, μοιραζόμαστε εμπειρία για τη δημιουργία ενός ε, Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ή Ινστιτούτου για την Ειρήνη. Κάτι το οποίο πολύ θέλει ο Υπουργός, ο πρόεδρος του Προπολογισμών. Υπέρ, παρακαλώ. Χωρί να θέλω να σα επηρεάσω βέβαια. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Η Φρανσίσα Μπράτνερ πρέπει να το μάθει αυτό, θα έρθει να με φιλήσει, λέει ο προεδρο 42 42-37, ανταλλαγή προγνωμένων. Υπό ηγητή, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51-85 της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Περισσότερο για περισσότερο, η αρχή δηλαδή αυτή. Συμφωνεί ο εισηγητής. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4276. Πρόθεση της μη βίας. Στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπληρώνει ο Πρόεδρος. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία υπέρ. Θα το ελέγξουμε. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 18 κατά συνεπώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την μη βία. 4102 ε, Δίκτυο υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι γελάτε, λέει ο πρόεδρος. Για μένα πρόκειται. Ο εισήγητης συμφωνεί, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44-14. Καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Ο εισηγητής συμφωνεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Να παληθεύσουμε ηλεκτρονικά γιατί κανένα χέρι δεν βλέπω να σηκώνεται. 44-14. Special focus on fight against antisemitism. Πέρα στις φοφορίες. Πέρα της 25 υπέρ 13 κατά εγκρίνεται. Καλύπτει και την επόμενη. Όχι, γιατί πρόκειται για διαφορετική γραμμή. 44-15. Συμφωνεί ο συγκεκριτής υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάλι είμαστε στην αρχή more for more. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία ALDE για το EUSBR project. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάλι πρόθεση της μη βίας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λέει ο Πρόεδρος. 4275. Κατά ο εισηγητής. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Με την ίδια πλειοψηφία που είχαμε και πριν για το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Λυκειωμένων υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Με την ίδια πλειοψηφία. Εξωτερικών υποθέσεων 50-62. Τώρα πάλι αρχή more for more. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα, 44-16, προσθέτοντας ε, πτυχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ελευθερία, θρησκείες κλπ. Υπέρ, υπέρ ουσίτης, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44-17, για το ίδιο θέμα. Με συγκητής συμφωνεί, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αν μπλόκα πρέπει να είχαμε ψηφίσει μαζί. Άλντε 84-41. Ο εισηγητής συμφωνεί. Δεσμεύσεις, οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε, δύο συν 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. αναπτυξη Ανάπτυξης 54-51. Υπάρχει προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Όχι. Παρακαλώ. Ναι. Θέλουμε να προσθεθεί η τροπολογία και να μην αντικαταστήσει το κείμενο, να είναι προσθήκη δηλαδή. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, πως η τροπολογία αυτή των ε, σοσιαλιστών είναι για να πρόκειται για προσθήκη και όχι για αντικατάσταση. Συμφωνείτε, κύριε Σιγητά, συμφωνείτε. Υπέρ, ποιο είναι υπέρ. Κατά ο Σιγητής βλέπω. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ως προσθήκη. Επόμενη τροπολογία πάλι της Αναπτυξιακής Επιτροπής. 5409. Κοινωνική προστασία. Υπέρ. Σιγητής, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τελευταία γραμμή. Τροπολογία σοσιαλιστών 8005. Έχουμε προφορική τροπολογία. Μετά από το capacity building, οικοδόμηση ικανοτήτων. Δεν ναι. Να το εξηγήσω γιατί στην αρχική τροπολογία μιλάει για την δημόσια δίκηση και για την ε, ε, τουρκοκυπριακή δίκηση, ενώ μπορεί να παρεξηγηθεί σαν να πρόκειται για την ε, τουρκική. Γι' αυτό κάναμε αυτήν ε, την αλλαγή εδώ και ελπίζω να ικανοποιήσει. Πράγματι, η διευκρίνηση αυτή είναι σημαντική, πιστεύω. Αλεξάνδρα Άλβαρο. Για να καταλάβουμε καλύτερα την τροπολογία, δεν θα μπορούσε να ερμηνευθεί με τον τρόπο με τον οποίο εμείς το βλέπουμε ότι αναγνωρίζεται δηλαδή και το τουρκικό τμήμα. Αν πείτε τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι σαν να αναγνωρίζετε ότι υπάρχει μια τουρκική κοινότητα. Όχι κοινότητα, εννοώ τον πληθυσμό, τον κόσμο. Αυτό εννοώ σαν κοινότητα, δεν εννοώ το κράτος. Όταν λέμε community εννοούμε την κοινότητα, του ανθρώπου δεν εννοούμε το κράτο, Αλλά βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπο να είναι πιο σαφέ. Πρόεδρος, εγώ σας προτείνω. Α, ο Γιάννη Μούλντερ πρώτα. Για να αποφύγουμε τη σύγχυση εδώ. Ίσως ε, τουρκόφωνη να πούμε, μήπως αυτό θα ήταν πιο ικανοποιητικό. Πρόεδρος. Είναι ένα λεπτό ζήτημα εδώ. Γιατί διπλωματικά σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνετε ότι οι λέξεις έχουν μεγάλη σημασία. Προτείνω λοιπόν να κρατήσουμε στην ψηφοφορία αυτή το εξή, ότι η τροπολογία αυτή απευθύνεται στο κατεχόμενο από τους Τούρκους τμήμα της Κύπρου. Αλλά χρησιμοποιούμε τη διπλωματική ορθή γλώσσα, που εγώ δεν γνωρίζω και σχετικά με την οποία προφανώς υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές εδώ σήμερα. Γι' αυτό θα ζητήσουμε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να μας δώσει τη σωστή διατύπωση. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Ότι μιλάμε για τους τυρκόφωνους στην ίσο της Αφροδίτης. Έλγα. Ναι, αλλά υπάρχει μια γραμμή προπολογισμού για ρογή στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Υπάρχει ήδη δηλαδή. Οπότε μπορούμε απλώς να το επαναλάβουμε εδώ. Αγγέλικα. Αυτή η γραμμή μιλάει για την τουρκική κοινότητα και όχι για την τουρκοκυπριακή ε, κοινότητα. Είναι 22.02.07.03 που έχω δουλέψει πάνω τα τελευταία χρόνια και θέλουμε να προσθέσουμε 3 εκατομμύρια που είναι εντάξει, αλλά εγώ ρωτάω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα χρήματα αυτά θα τα δώσει πού για, στην Επιτροπή για τους Αγνοούμενους και πόσα στην ε, Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Ελπίζω η Επιτροπή να απαντήσει κάποια στιγμή, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Εδώ πρόκειται για μια ρύθμιση που έχει πολιτική έκφραση αν αλλάξει αυτό. Εγώ Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να ξέρουμε ότι αν αλλάξουμε το πολιτικό μήνυμα της ρύθμισης, δεν είναι μια καλή εικόνα που θα στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό προσωπικά σας ζητώ να το σκεφτείτε. Καλώς, Αγγέλικα. Ευχαριστούμε. Μην μπούμε τώρα στη συζήτηση επί της ουσίας. Υπάρχει πρόταση του Αντιπρόεδρου Καλφίν να αναβάλουμε για αύριο την ψηφοφορία αυτή, αφού επαληθεύσουμε προηγουμένω και διευκρινίσουμε το κείμενο πώς πρέπει να έχει. Συμφωνεί, καλώς. Η πρόταση αυτή λοιπόν, πολύ σωστή, του κύριου Καλφίν, μας οδηγεί στην λήξη των εργασιών μας για σήμερα. Συνεπώς, συνεπώς σας ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα όσους μέχρι το τέλος είχαν την υπομονή και ψήφιζαν. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ επίσης όλους τους συνεργάτες, τη γραμματεία, τους συνεργάτες των ομάδων, τους βοηθούς των μελών για την εξαίρετη δουλειά που έχουν κάνει και μας διευκόλυσαν το δικό μας έργο ώστε να επιταχυθεί η ψηφοφορία. Στόχος μας τώρα είναι να ολοκληρώσουμε αύριο το πρωί και να μην χρειαστεί να έρθουμε πάλι αύριο το απόγευμα. Στόχος είναι αυτός. Δεν είναι απόφαση, στόχος είναι. Συμφωνεί. Συνεπώς, διακόπτουμε. Προτείνω στους συντονιστές και τους βοηθούς τους να παραμείνουν στην αίθουσα. Χρειαζόμαστε τον εισηγητή με τους συντονιστές. Όχι, όχι. Συνεπώς διακόπτουμε πέντε λεπτά και συνεχίζουμε με τους συντονιστές. Έληξε συνεδρίαση.